Καλημέρα σας. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της θεσινής συνεδρίας έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσεις. Όχι. Θεωρούνται λοιπόν εγκεκριμένα. Έχω επίσης μια ανακοίνωση να σας κάνω. Έχω λάβει από την